κυριών Dodge, Ford, του κυρίου Καν και του κυρίου Λούερ στα εθνικά τους κοινοβούλια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταγράφει την γενότητα της θέσης τους από τις 9 Ιουνίου 2017 σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό. Οι αρμόδιες αρχές της ε, Δημοκρατίας της Πορτογαλίας